πρέπει να ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, πάντα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να έρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο όπου έχω διατελέσει μέλος δύο φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα κοινοβούλιο ε, το οποίο γνωρίζω και χαιρετίζω τον ουσιώδη πολιτικό ρόλο. Προετοιμάζομαι για τα καθήκοντά μου ως Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνίων στην Επιτροπή του Ζαν claude Juncker. Και το πράτο με υπερηφάνεια, την υπερηφάνεια εκείνου που ετοιμάζεται να υπηρετήσει το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Προετοιμάζουμε με ταπεινότητα και κυρίως με το αίσθημα μιας τεράστιας ευθύνης απέναντι στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που καλούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Έχω μια βαθιά πολιτική πεποίθηση εμείς είμαστε η Ευρώπη της τελευταίας ευκαιρίας. Αυτή την πεποίθηση την έχω σφυριλατήσει κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας όπου τα ευρωπαϊκά ζητήματα ήταν πάντα στο προσκήνιο. Διετέλεσα Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου σας, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και τέλος τα δύο τελευταία έτη ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας. Από όλη μου την ιστορία και με κάθε ικμάδα μου είμαι βαθύτατα Ευρωπαίος. Η Ευρώπη στα μάτια μου είναι η μεγάλη πολιτική εποποιία, επιτρέψτε μου να το πω, του αιώνα μας. Πιστεύω βαθύτατα ότι οι διαφορές μας μας πλουτίζουν, ότι η προσέγγιση των λαών είναι από μόνη της αξία, ότι είμαστε πιο δυνατοί όταν μιλούμε με μία φωνή. Είμαι πεπισμένος ότι η ευρωπαϊκή ιδέα μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε το τραγικό παρελθόν της Υπήρου. Αυτό τον καιρό παντού στην Ευρώπη ε, ε τιμούμε την επέτειο των 100 ε, ετών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα 70 χρόνια από την ναζιστική βαρβάρια και συγγνώμη. Η Ευρώπη γεννήθηκε για να βγει από το χάος, θυμόμαστε, και το χάος χτυπάει την πόρτα μας. Ε, οι ρίζες μου είναι πολωνικές από τη μητέρα μου και ρουμανικές από τον πατέρα μου. Είμαι από μια οικογένεια που έζησε τις περιπλανήσεις του κόσμου του χθε. Ε, για το οποίο μιλούσε ο Στέφαν Τσβάικ και ε, που γνώρισε την τρομακτική ε, τραγωδία, την απίθμενη τραγωδία του ολοκαυτώματος. Είμαι πεπισμένος ότι η επανένωση της Υπήρου μας το 2004 και συνέχεια στο 2007, όπου συνεισέφερα ως εισηγητής για την προσχώρηση της Ρουμανίας, χώρα όπου γεννήθηκε ο πατέρας μου, ήταν ιστορική στιγμή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Με δύο λόγια, για μένα έχει πολύ βαθιά πολιτική σημασία το να είναι κανείς πρωταγωνιστής στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα και χτες και σήμερα. Και έχω και μια προσωπική σχέση με αυτό. Ξέρω ότι είναι όλο και πιο λίγοι πολίτες που έχουν αυτό το όραμα σήμερα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι αυτονόητη η Ευρώπη για όλους. Πολλοί πολίτες σήμερα είναι απογοητευμένοι γιατί πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν κατάφερε να τους ε, προστατεύσει και να ε, προχωρήσει στις απαραίτητες πρόοδους ότι είναι ανεποτελεσματική πολιτικά και ανίκανη οικονομικά. Αυτό το βλέπω να ενισχύεται ως αίσθημα ε, και στα λαϊκά στρώματα και στους ε, εργάτες. Και δεν ε, είμαι διατεθειμένος να το δεχθώ αυτό ως πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα πρέπει να σταματήσουμε να ζητούμε από τους Ευρωπαίους να κάνουν υπομονή. Τους νέους, τους πιο ηλικιωμένους, τις γυναίκες, τους άντρες, παντού που ανησυχούν. Δεν μπορούμε να τους απαντούμε ότι έχουμε ειρήνη στην Ευρώπη και συμφιλίωση ε, από τους χθεσινούς εχθρούς έχουμε σήμερα φίλους στην Ευρώπη. Θα πρέπει να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο, με αποτελέσματα και με τη βοήθειά σας θέλω πλήρως να συνεισφέρω σε αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε με την πλευρά ε, της ελπίδας και της πολιτικής βούλησης. Παραστάτες και αυτό είναι το μήνυμά μου και θα το διατηρήσω καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Η Ευρώπη έχει κάνει πρόοδο στα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι τη συγκίνηση που νιώσαμε εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έγινε η διεύρυνση το 2004. Θυμάμαι πιο πρόσφατα στο Eurogroup και στο ECOFIN τα δύο τελευταία χρόνια τις μακρές νύχτες. Ήταν μια πραγματική υπαρξιακή αμφιβολία αυτή που πλανόταν στην Ευρώπη. Και ε, κάθε εβδομάδα συναντιόμαστε για να αποφύγουμε την καταστροφή και την έκρηξη της Ευρωζώνης και την ε, χρεοκοπία των τραπεζιών. Με την ε, πολύτιμη κομβική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, σταμάτησαν ε, οι κερδοσκόποι να ποντάρουν στη διάλυση της Ευρωζώνης. Οι χώρες που είναι σε προγράμματα έχουν θυσίες υποστεί και μάλιστα επώδυνες. Έχει μπει σε μια τροχιά η Τραπεζική Ένωση ε, και τα δημόσια ελλείμματα έχουν μειωθεί. Έχω σημειώσει ε, και εγώ ε, τη συμμετοχή μου σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να χρειάζεται οπωσδήποτε οικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα, αλλά οι πολίτες κυρίως τι ζητούν. Κοινωνική πρόοδο, ανάπτυξη, απασχόληση. Η πρόκληση είναι να αγωνιστούμε όλοι για να μην ε, έρθει οικονομική κατάπτωση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εξορκίσουμε αυτή την απειλή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα είμαι ευτυχής που έχω την ευκαιρία να ε, εργάζομαι και να υπηρετώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δημόσιο Συμφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μαζί με το Κοινοβούλιο είναι η ουσιαστική καρδιά αυτής της υπόθεσης και ε, αισθάνομαι έτοιμος. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ το συζήτησα αυτό με τον πρόεδρο Ιούνκερ και χαίρομαι ε, που θα έχω την ευκαιρία να μπω στην ομάδα του. Ε, θέλω να συνεργαστώ απολύτως με τους συναδέλφους μου, αντιπροέδρους, επιτρόπους. Γιατί θα πρέπει η κοινή ευφυΐα και αποφασιστικότητα του καθενός να μας βοηθήσουν για να βγάλουμε την Ευρώπη από τη σημερινή κρίση στη θέση που μου αναλογεί και με το συλλογικό πνεύμα που καθιστά την Ευρώπη μοναδική ως δύναμη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω εδώ να χαιρετήσω ε, τους κυρίους όλοι, Ρεν και, το, και σε μετά και τον Μισελ Μπαρνιέ ε, με τους οποίους συνεργάστηκα για την Τραπεζική Ένωση από τα προηγούμενα καθήκοντά μου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά μπροστά μας και θέλω να ε, προχωρήσουμε με την πολιτική και δημοκρατική συνδρομή του Κοινοβουλίου. Θα συνεργαστούμε την επόμενη πενταετία και ε, το φύλλο πορεία μας, ο δικός χάρτης είναι πολύ σημαντικός και απαιτητικός. Θα πρέπει η οικονομία να ξανασταθεί στα πόδια της των πολιτών και των επιχειρήσεων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, μία σαφή πορεία να χαράξουμε. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Είναι διπλή αυτή η προσπάθεια και αποφασιστική η μάχη. Από τη μια θα πρέπει να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της οικονομίας μας και από την άλλη ε, να έχουμε την ανάπτυξη. Αυτά είναι δύο βασικές συντεταγμένες και δεν θα πρέπει να τις φέρνουμε αντιμέτωπες. Να σταματήσουμε τις πολιτικές διαφορές, τις προσωπικές επιθέσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν νοείται ε, ανάπτυξη χωρίς τη μείωση του χρέους, ιδιωτικού και δημοσίου. Δεν νοείται μείωση του χρέους όμως και ε, πρόοδος χωρίς ανάπτυξη. Είναι αλληλένδετα και δεσμεύομαι λοιπόν εδώ ενώπιόν σας να ε, επιβάλλω το σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη. Χωρίς συγκατάβαση και χωρίς υπερβολική αυστηρότητα. Θα πρέπει όλες οι χώρες, μεγάλες ή μικρές, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση βάσει της αξίας και των ίδιων κανόνων θα πρέπει ε, να σας πω ότι θα είμαι ένας διαιτητής δίκαιος και αμερόληπτος. Μπορείτε να υπολογίζετε σε αυτό. Έτσι ώστε όλοι οι πάντες, όποιος και είναι αυτός, οποιοδήποτε, να παίζει με τους ίδιους κανόνες στην οικονομία μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ξαναδούμε το μείγμα πολιτικής στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενίσχυση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, αναθεώρηση στρατηγικής του 2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει ανακοινώσει ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ. Αυτό είναι μια ευκαιρία για να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Είμαι δεσμευμένο επίση και προσιλωμένο στην ενίσχυση τη Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει και εμβάθυνση τη πολιτική και θεσμική αρχιτεκτονική, τη λειτουργία των μέσων, αλλά και συνέχιση τη διεύρυνση προ άλλα κράτη-μέλη που θα πληρούν τα κριτήρια αγωνίστηκα σκληρά για να ε, εξασφαλίσουμε το ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θα συνεχίσω να το πράττω αυτό χέρι με χέρι με το Βάλτις Ντομπρόφσκης, διότι πιστεύουμε βαθύτατα στο μέλλον του κοινού μας νομίσματος. Επίσης, δεσμεύομαι ενώπιόν σας να εργαστώ σκληρά για να επανέλθει η ανάπτυξη. Δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται ε, να δεχτούμε άλλο ένα σενάριο μηδενικής ανάπτυξης για το επόμενο έτος. Έξι χρόνια μετά την αρχή της ε, κρίσης, ε, οι επενδύσεις στην Ένωση συνολικές είναι κατά 17% χαμηλότερες στο επίπεδο του 2007. Θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου για το αναπτυξιακό σχέδιο των 300 δισεκατομμυρίων που ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ εδώ ανακοίνωσε. Επιγόντως χρειάζεται η Ευρώπη επενδύσεις και ιδιωτικές και δημόσιε. για νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, υποδομές που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Θα εργαστώ σκληρά τους επόμενους μήνες για το στόχο αυτό μαζί με τον Γέρκη Κατάινεν και τον Τζόναθαν Χιλ. Επίσης ελπίζω ότι η ανάκαμψη θα φέρει και μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη για τους πολίτες μας. Θα πρέπει να διορθώσουμε τις ζημίες που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση, που έχει προκαλέσει τόσα πολλά δεινά στους άνδρες και τις γυναίκες παντού στην Ήπειρό μας εδώ και πάλι δεν επιτρέπεται και δεν θα έπρεπε να δεχθούμε επίπεδα ανεργίας που φτάνουν στο 11,2% στην Ευρωζώνη και ε, εκτοξεύονται στο 23,3% για τους νέους μας. Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η φόρος, να δημιουργεί ε, τις θέσεις εργασίας του αύριο, να ξαναδώσει την εμπιστοσύνη στους νέους Ευρώπης. Σε αυτό το θέμα έχουμε ε, συναντήληψη με τη Μαριάν Τάισεν φέρω μαζί μου αυτή την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη αλλά επίσης ε, έχω και την ευθύνη της ε, ε, φορολογικής πολιτικής. Εδώ θα συνεχίσω ε, τον αγώνα κατά των φορολογικών παραδείσων της φοροαποφυγής και της επιθετικής ε, φορολογικής πολιτικής και σχεδιασμού. Αυτό είναι σημαντικό και για οικονομικούς και για δεοντολογικούς και ηθικούς λόγους. Τερματίσαμε το τραπεζικό απόρριτο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Όπως αποφάσισε το G20, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει στην Ευρώπη να γίνει κανόνας και σε παγκόσμιο επίπεδο προδιαγραφή και πρότυπο και ε, να είστε βέβαιοι ότι θα σας υποστηρίξω σε αυτή την κοινή μας μάχη. Επίσης θα βοηθήσω τα 11 κράτη-μέλη που αποφάσισαν να δημιουργήσουν και να θεσπίσουν ένα ε, φόρο επί των χρήματο πιστοτικών συναλλαγών. Ε, αυτή την ε, πρωτοβουλία την υποστήριξα από την αρχή μαζί με τον Wolfgang Schäuble και θα συνεχίσω να το πράττω ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ας μην λησμονούμε και τα τελωνιακά ζητήματα που αφορούν πολύ συγκεκριμένα θέματα για την προστασία των πολιτών μας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μα σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Θα πρέπει από κοινού να εργαστούμε για να τεθεί σε ισχύ ο νέος τελωνιακός κώδικας μέχρι το Μάιο του 2016. Είναι κομβική αυτή η ευθύνη, θα συνεργαστώ πολύ στενά με τα μέλη της Επιτροπής ΙΜΚΟ και ΙΝΤΑ. Ιδού λοιπόν ορισμένα από τα θέματα που προετοιμάζομαι να επομιστώ ε, με τη βοήθειά σας. Ο Ζαν Κλωτ Ιούνκερ θέλει σε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο αποτελεσματική, πιο πολιτική, πιο συνεκτική. Εκεί θέλω να είμαι αγγιητής του ευρωπαϊκού συμφέροντος το πω αλλιώ και καλύτερα του ευρωπαϊκού οικονομικού συμφέροντος. Ε, ο άγρυπνος θεματοφύλακας των κοινών κανόνων. Γνωρίζω ε, ότι κάποιοι προβληματίζεστε. Είμαι Γάλλος, είμαι σοσιαλδημοκράτης, ε, πώς να το αρνηθεί κανείς. Ε, το λέω ανερυθρίαστα. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν θα είμαι πρέσβης μιας χώρας ή ενός κόμματος. Όπως είστε σε θέση και έχετε ε, το δικαίωμα και δίκιο να απαιτείτε, θα είμαι απολύτως ανεξάρτητος, αμερόληπτος απέναντι σε κάθε συμφέρον, ιδιωτικό ή εθνικό. Στο πλευρό σας θέλω να υπηρετήσω την ευρωπαϊκή υπόθεση. Είπα ότι είμαστε η Ευρώπη της τελευταίας ευκαιρίας. Το πιστεύω, είμαι ακράδαντα πεπισμένος. Η Ευρώπη είναι ένα θαυμάσιο πολιτικό εγχείρημα. Και όπως όλα τα πολιτικά εγχείρηματα, ε, έχει και αδυναμίες, ε, είναι και θνητή. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου θα είμαι πάντα πρόθυμος να συνεργάζομαι με το Κοινοβούλιο, με όλους σας, όλους εσάς και στις ομάδες σας. Και προσβλέπω ε, στις δύο γενικές διευθύνσεις ε, για τη βοήθειά τους. Πάντα με διάλογο, ε, αφού στο Κοινοβούλιο. Έχω μεγάλο σεβασμό για το Κοινοβούλιο που το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής και πάρα πολύ περήφανος ως Ευρωβουλευτής. Έχουμε εμπειρία και εγώ έχω μακρά πείρα και ευρωπαϊκή και εθνική και ξέρω πώς η δημοκρατική ευθύνη είναι σημαντική για τα θεσμικά όργανα. Αυτά όλα θα με διέπουν στη δράση μου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα είμαι ένας επίτροπος υπεύθυνο και έχοντας πάντα υπόψη αυτή τη δημοκρατική δέσμευση. Ζητώ σήμερα την υποστήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας αναμένουν σε αυτό το πνεύμα και με ειλικρίνεια θα απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις, όποιες και είναι αυτές. Σας ευχαριστώ.